Πρώτη έκθεση είναι η έκθεση Φεράρα σχετικά με την αίτηση, ασυλία, αίτηση για την άρση της ασυλίας της Μαρίν Λεπέν. Έχει κατατεθεί πρόταση από τον κύριο Κόρβιν, Μίκε για την αναβολή της σχετικής ψηφοφορίας. Σύμφωνα με τον κανονισμό, όπως με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου, αυτή η πρόταση για να γίνει αποδεκτή πρέπει να κατατεθεί εξ ονόματος μιας πολιτικής ομάδας. Πράγμα που δεν ισχύει στην περίπτωση του κυρίου Κόρβιν Μίκε, ο οποίος είναι μη εγγεγραμμένος. Και με την ευκαιρία επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό άρθρο 180 παράγραφος 1 η ψηφοφορία για αιτήσει άρση της ασυλίας οποιοδήποτε ευρωβουλευτή γίνονται με απλή ψηφοφορία. Επομένως, προχωρώ στην ψηφοφορία πώς είναι υπέρ της άρσης της ασυλίας. Κατά αποχές η ψηφοφορία είναι σαφής, εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στην έκθεση Μανέσκου. Προχωρούμε στην έκθεση Μανέσκου για τη σύνδεση παρακαλώ μη φωνασκείτε να εμπιστεύεστε και το Προεδρείο και τα μάτια σας. Ήταν συντριπτική η πλειοψηφία. Προχωρούμε στην έκθεση Μανέσκου για τη σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβάνου σε ό,τι αφορά στην προσχώρηση της Κροατίας. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προχωρούμε στην έκθεση Βάιντεν Χόλτσερ. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προχωράμε στην έκθεση Κράσνο-Τέψικη. Τροπολογία 51. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, που σημαίνει ότι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου περατώθηκε. Η επόμενη αφορά υποχρεώσει στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων. Ψηφοφορία με ανάταση της χειρός. Όσοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προχωρούμε στην έκθεση Καμπεθόν Ρουίς. Υπάρχει τροπολογία 1 με ανάταση της χειρός. Όσοι είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 8 ψηφοφορία μονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 22 του αρχικού κειμένου με ανάταση της χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 θα κάνουμε ευχαρίστως έλεγχο για την παράγραφο 22 του αρχικού κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. Ε, Παράγραφος 50, τροπολογία 2 από 76, πάνω από 76 συναδέλφους. Με ανάταση της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κάνουμε έλεγχο για την τροπολογία 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Με ανάταση της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59. Ήταν σαφές. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο για την τροπολογία 3. Κάνουμε έλεγχο. Βεβαίως Βεβαίως, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 3. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η, τροπολογι η παράγραφος 59 σε δύο μέρη με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά αποχές θα χρειαστεί έλεγχος για το δεύτερο μέρος με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Με ανάταση της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 95 του αρχικού κειμένου. Όχι, απορρίπτεται καθαρά. Η παράγραφος 95 του αρχικού κειμένου. Συγγνώμη, εγκρίνεται, συγγνώμη, εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 95 του αρχικού κειμένου. Με ανάταση της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η παράγραφος 98 του αρχικού κειμένου. Όχι, ήταν καθαρή η, διαφορά. Η παράγραφος 98 του αρχικού κειμένου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφοφορία στο σύνολο του κειμένου νομονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνούμε στην έκθεση Κώστα. Τροπολογία 8 με ανάταση της χειρός. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η παράγραφος 1 του αρχικού κειμένου με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά Παρακαλώ μη φωνασκείτε, είναι μεγάλη η διαφορά. Απορρίπτεται με συντριπτική πλειοψηφία. Μην καθυστερούμε για φανερά αποτελέσματα. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 45 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 ψηφοφορία με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 21 επίσης με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται επίσης. Τροπολογία 1. Με ονομαστική κλίση υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη γ, τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο στην αιτιολογική σκέψη ΙΓ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 στην αιτιολογική σκέψη ΙΕ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία, ε, ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Yeah. Ο, ο κύριος Πρέντα. Κύριε Πρόεδρε, μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού unblock όλες τις τροπολογίες που αφορούν της ομάδας, της ομάδας Λεπέν. Παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω μεγάλη εκτίμηση στην διεύθυνση, αλλά παραβιάζεται την αρχή της ισότητας. Πρώτον, δεν κοιτάτε καν πώς είναι η ψηφοφορία. Αγνοείτε όσους ζητούν point of order. Εκτιμώ λοιπόν τη διεύθυνση της συζητήσεως, αλλά θα πρέπει να είναι δημοκρατική και δίκαιη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ομπερμπάγκερ για την εκτίμηση που δείχνετε στον Προεδρεύοντα και στους συνεργάτες του. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι όλες οι ψηφοφορίες που έγιναν με ανάταση της χειρός είχαν πολύ σαφές αποτέλεσμα. Οι τροπολογίες πολιτικής ομάδας απορρίφθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία και αυτό φάνηκε και στις ψηφοφορίες που ζητήσατε να γίνουν με roll call vote. Ήταν η ίδια συντριπτική πλειοψηφία που τις απέρριψε. Τώρα σε, ο, ε, θέλει επίσης η κυρία Κώστα, ο το Πρόεδρε, να πω ότι σήμερα είναι σημαντική μέρα, γιατί το Κοινοβούλιο αποφάσισε να στηρίξει και άλλο τον πολιτισμό που τον χρειαζόμαστε στην Ευρώπη, γιατί δημιουργεί αξία ε, και πολιτιστική, ε, πολιτιστικό πλούτο και προσφέρει δουλειά στους νέους. Δυστυχώ, ε, δεν λειτουργήσε το μηχάνημά μου και δεν μέτρησε τη θετική μου ψήφο τη στιγμή τη ψηφοφορία. Ήθελα να το πω, τραγική ηρωνία. Ήθελα να καταγραφεί ότι ψήφισα υπέρ. Η διευκρίνησή σα θα ληφθεί υπόψη. Τώρα προχωρούμε στην έκθεση Χιμένε Μπαρμπάτ και θέλω να πω, όπως με ενημερώνουν και οι συνεργάτε μου για την πρόταση του κυρίου Πρέντα, ότι μπορούμε να ψηφίζουμε τροπολογίες unblock μόνο όταν είναι συναφές και συμβατό το περιεχόμενό του. Επομένω, ω Πρόεδρος που οφείλω να τηρώ τον κανονισμό, δεν μπορώ να εθετήσω την πρόταση του κυρίου Πρέντα. Προχωρούμε με μια διαδικασία σφιχτή στην ψηφοφορία όπως έχει οριστεί. Τροπολογία 12 με ανάταση τη χειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφοφορία στο σύνολο του κειμένου μονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Λήξη ψηφοφορίας. Η έκθεση εγκρίνεται. Προχωρούμε στην τελευταία έκθεση του κυρίου Μακλάρκιν. Τροπολογία 1. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση για το σύνολο του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Προχωρούμε σε αιτιολογήσεις ψήφου.